Good morning, colleagues. I am happy to announce that this meeting... Καλημέρα, συνάδελφοι. σας αναγγέλω ότι θα αρχίσει η συνεδρίασή μας. Οπότε καθίστε για να αρχίσουμε. Σήμερα οι χαιρετισμένοι είναι οι σοσιαλιστές γιατί είναι εδώ. Έχουν κάτσει και περιμένουν να ξεκινήσουμε. Οπότε εσείς είσαστε πρωταθλητές σήμερα. Και ακριβώς αυτό θα πω στο ΕΛΚ. Καλά, καλά, πλάκα σας κάνω. Οπότε όποιο είναι εδώ, τα έμαθε ποιο δεν είναι, δεν τα ξέρει αυτό. Για να δούμε τώρα τι αποφάσισαν χθε οι συντονιστέ. Έχουμε την, το σχέδιο τη διάθεση για τον Ιούνιο, έχουμε τι ε, εκθέσει και τι νομοδοτήσει και με χαρά μου σα αναγγέλω ότι ο Νότης μαριά ο συνάδελφο από το ECR, είναι ο εισηγητή τη νομοδότηση όσον αφορά την διασυνοριακή ε, αναγνώριση των ε, υιοθετήσεων για την Γιούρη που είναι η αρμόδια ε, Επιτροπή. Και επίσης είπαμε στην ε, γραμματεία μας να συνεργαστεί για αυτό το λόγο με την γραμματεία της Γιούρη, ούτως ώστε αυτό το εργαστήρι να προετοιμαστεί. Είναι αυτό το οποίο το επιθυμούσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση και θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή σχετικά με αυτή τώρα όσον αφορά τα κατεπήγοντα και ε, αυτά τα οποία έχουν ζητήσει οι πολιτικές ομάδες. Επίσης, συμφωνήσαν χθε οι συντονιστέ όσον αφορά την ε, αναφορά 1772 κάθετος 12 και άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα, δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν κλαπεί στην Ισπανία, όλα αυτά να μπουν στην ε, ε διάταξη τον Σεπτέμβριο. Για την θαλεδομίδη επίσης στην Ισπανία και αυτό θα μπει στην μέση διάταξη τον ε, Ιούλιο φέτος. Επίσης έχουμε κάποιες ερευνητικές ε, αποστολές και αποφασίσαμε να κάνουμε μια αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος. Φέτος, το δεύτερο εξάμεινο του 2015, τώρα όσον αφορά τα θέματα προστασίας των ανηλίκων. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια ερευνητική ε, αποστολή αρχάς του 2016 στην Ισπανία. Και αυτό θα αφορά κυρίως τις ε, αναφορές όσον αφορά τον ποταμό Εύρο και τον ποταμό Τάχο για τα θέματα διαχείρισης ε, τα συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Τώρα, σε συνέχεια, έχουμε κάποιες αναφορές για κάποιες ε, απατηλές ε, πρακτικές της Πανικής Τράπεζας και είπαμε ότι θα απευθυνθούμε στην διάσκεψη των Προέδρων και κατά αυτόν τον τρόπο αυτό να ενταχθεί στην ημέρη διάταξη της Ολομέλειας οπότε θα υπάρξει κάποια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια για αυτό το θέμα των τραπεζών. Ε, δεν ξέρουμε αν θα εγκριθεί αυτό, αλλά πάντως πρόθεσή μας είναι να καταθέσουν αυτό το αίτημα. Οπότε θα υποβληθεί για ψήφιση τον Ιούνιο στην Επιτροπή. Επίσης αποφασίσαμε να υπάρξει μια επιστολή την οποία θα στείλουμε ε, στον φορέα των τραπεζών στην Ισπανία. Η ε, διαδικτυακή πύλη τώρα. Είπαμε η επικεφαλής η μας εδώ να ασχοληθεί με αυτό και ο συνάδελφος εδώ επίσης ήταν εκεί και το συζητήσαμε και το πήγε πάρα πολύ καλά η γραμματεία μας μέχρι τώρα. Επίσης αποφασίστηκε η κυρία Ρώσα Στάρας από το ΕΛΚ να μας εκπροσωπήσει στην ομάδα εργασίας της Γιούρ για το Διοικητικό Δίκαιο και επίσης κάποιος από τους φιλελεύθερους πρόκειται να είναι αναπληρωτής εκεί. Θα βρούμε ποιος είναι. Τι άλλο έγινε. Α, ναι. Έχουμε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές. Εκείνες οι οποίες έχουν διανεμηθεί. Πρόκειται για ένα μεγάλο έγγραφο και αποφασίστηκε οι συντονιστές να υποβάλουν τις απόψεις τους ή τις τροπολογίες τους εγγράφος μέχρι τις 28 Πέμπτου στην γραμματεία. Η γραμματεία έχει πια τα έγγραφα, δεν τα έχω και το πρώτο θέμα θα ζητηθεί από τους συντονιστές τον Ιούνιο. Οπότε θα έχουμε τις νέες κατευθυντήριες που θα εγκριθούν στην συνεδρίαση του Ιουλίου πριν τις σερινές διακοπές. Και τώρα. Αυτά από τους συντονιστές. Μάργαρετ, έχεις το λόγο. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να μην και χθε. Μου είπαν ότι για την διευθυντική αποστολή επίση αποφασίσαμε να πάμε στην Ιρλανδία. Το έχουμε υποσχεθεί εδώ και καιρό. Συμφωνώ πολύ με την Ισπανία, αλλά έχουμε πάει πολλέ φορέ εκεί. Καλό θα ήταν να επιμείνουμε στην αποφασή μας και να πάμε στην Ιρλανδία. Αυτά μου είπαν για τις αποφάσεις χθε. Πρόεδρος, ναι, το συζητήσαμε επί μακρόν και αυτό θα κάνουμε μάλλον το 2016. Ναι, επισήμω δεν πήραμε την απόφαση. Ας πάρουμε την απόφαση στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Αν με επιτρέπετε, για να το ξεκαθαρίσω. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση για την Ιρλανδία θα πάρουμε αυτή την απόφαση. Αλλά είχαμε δύο αποφάσεις. Μία για το 2015 Ηνωμένο Βασίλειο, 2016 Ισπανία. Και μάλλον θα γίνει και διαρευνητική αποστολή και στην Ιρλανδία. Αλλά δεν έχει αποφασιστεί επισήμω. Ωραία, μπορούμε τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες.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 έχουμε την ε, συνέχιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ε, Πολιτών Right to Water. Κυρία Όκεν είναι η συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα έχω την ε, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά. Α, ναι, ένα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβουλευτική α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβουλευτική τοπολογία β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τοπολογία 3, υπέρ, Α, ναι, καταπληκτή, βεβαίω. Είναι νωρί, ξέρετε. Έχω ξυπνήσει νωρί σήμερα. Τροπολογία 4 κατά 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλησπέρας. Απορρίπτεται. Β' τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Θέλατε να ελέγξουμε, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η επόμενη. Περνάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7 καταπληκτή, Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. καταπληκτή. Πάμε στη 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές να τα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Ασυμβαστική δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Καταπίπτει. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να τα ελέγξουμε. Άρχιτε ψηφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. 21 υπέρ. Α, και αυτή καταπίπτει. 24. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί 22, 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25, κατά περίπτωση 26, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Α, όχι. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 καταπίπτει και 43. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, α, όχι, καταπίπτει. 54 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό τη. Ελεκτρονικά θα ψηφίσουμε βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, ψηφίσατε πολύ. Από το EFTD έχουμε δύο παραπάνω. Λοιπόν, να κλείσουμε την ψηφοφορία και να την επαναλάβουμε. Οι συντονιστές να ελέγξουν ότι έχουν επαρκή αριθμό μελών και όχι παραπάνω. Άρχεται ψηφοφορία. Και πάλι. Αυτό η FTD είστε παραπάνω. Ένας παραπάνω. Και από τους σοσιαλιστές επίσης ένας παραπάνω. Α, δύο παραπάνω έχετε το FTD.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 28 ψηφίσαντες, πέρας ψηφοφορίας. And Λοιπόν, εγκρίθηκε με ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Excellent work. Εξαιρετική δουλειά. that was strange. That was a bit strange. Okay. Now the application of EU law. Here we are. Let's proceed to the, the second vote. Να περάσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Για την ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού ε, Νόμου. Ο συνάδελφος ε, Ρώσα. Προπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. The vote is open. Έλεγχος παρακαλώ. Again, check that you have the sufficient... Ελέγξτε αν έχετε επαρκείς ε, ψήφους. Πέρας ψηφοφορίας. Έγκρινε Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 11. Σε δύο διαφορετικές εκδοχέ, Η πρώτη εκδοχή υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης συγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξω γιατί δεν σηκώνουν τα χέρια. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 12 ηλεκτρονικά. Τι 12. Πέρας ψηφοφορία τώρα. Με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται εσά. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας, Ιτάλος. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Μα τα σηκώνει ο κόσμος τα χέρια του. Η 13 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές Έγκρινεται. Η 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. άποχέ, Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει 25 λοιπόν τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορίας για την 32. And it's closed. Εγκρίνεται. Μα, δεν έχει μεγάλη φορά, αλλά παρόλα αυτά εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ωραία. Ας ελέγξουμε την 37. έξι ψηφοφορίας παρακαλώ. Πάλι υπερισσεύουν ψήφοι. Συντονιστέ, παρακαλώ, προσέξτε να μην έχετε πολλέ ψήφου. Ωραία, τώρα είμαστε οκ. Okay. Ένδοξη ψηφοφορία, πέρα. Εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά. Η 38 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος λοιπόν, εντάξει. Έναξη ψηφοφορία. Την 38 ψηφίζουμε. Την 38. Περισσεύει μία ψήφος. If this machine is not completely... Okay. Αν δεν κάνει λάθος το μηχάνημα. Πέρας ψηφοφορίας. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει ισοψηφία, απορρίπτεται. Το ξέρω, το ξέρω. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε, έστω, έστω, ας το ελέγξουμε. Έναξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία υπερθμό 40. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Σε υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται σαφέστατα. 46 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, επίσης εγκρίνεται. Technical issues, I guess. Okay, can I proceed? Okay, okay. So, amendment Η 48 στην πρώτη της εκδοχή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 48 the version 1. 48 πρώτη εκδοχή παρακαλώ να ψηφίσουμε. Mm. Έναρξη ακόμα τη ψηφορία, Τώρα πέρασε. Εγκρίνεται. Uh, Και έτσι λοιπόν η δεύτερη εκδοχή καταπίπτει. Και περνάμε λοιπόν κατευθείαν στην 4. Υπέρ. Συμβαστική 4. Υπέρ. Συμβιβαστική 4 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. 53, the vote. Την 53 έναρξη. And the vote is now closed. And it is. Πέρα. 54 in favor. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 55. 50, 54. 54 παρακαλώ. Ας ελέγξουμε. The vote is open. And now it's closed. Πέρας τη φορία. Απορρίπτεται. By one vote. But we, I need to check all the time. I, I realize that. 55 in favor. 55 υπέρ. έχει. Abstentions clearly carried. 50... Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Yeah. Because you raised your hand for a yes. Okay, let's, let's, let's take it once more. 56. Πάμε πάλι. 56 υπέρ α Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι σαφές. Ε, τώρα εντάξει. Πείτε, σηκώστε το χέρι σας όπως έπρεπε. Ναι, ναι, ναι, Μάλλον τη στιγμή που θέλετε ήταν σαφές. Τεχνικό διάλειμμα. But what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 Πλήρη σύγχυση. Πλήρη σύγχυση. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην 49, λέει πρόεδρο, γιατί το δεύτερο τμήμα κατέπεσε. Και τώρα σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 49, την οποία και δεν ψηφίσαμε. Το πρώτο τμήμα μόνο εγκρίθηκε. Να πάμε στην 49, λοιπόν, σα παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, περνάμε στην τροπολογία 56. Υπέρ. Α, ψηφίσαμε την 56, λέει η πρόεδρο, στην 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν τώρα ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία. Α, Πίτερ, Δεν ξέρω. Αν δεν κάνω λάθος, στην τροπολογία 11 έχουμε, είχαμε και εκεί δύο εκδοχές. Στην 11, 11. Και ψηφίσαμε υπέρ και των δύο εκδοχών. Είναι δυνατόν ή ε, μήπω θα πρέπει να καταπέσει η δεύτερη, αν έχουμε υπερψηφίσει την πρώτη. Το ρωτάω, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν έχουμε υπερψηφίσει την πρώτη εκδοχή, πώ γίνεται να εγκριθεί και η δεύτερη μετά. The second fall, or I don't know. Δεν πρέπει να καταπίπτει η δεύτερη εκδοχή. Πριν ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου. Exactly. The first... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Η πρώτη εκδοχή υπερψηφίστηκε. Αυτό σημαίνει ότι καταπίπτει η δεύτερη εκδοχή. It was also voted, but the consequence is that it's false. Ναι, αλλά καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. Έχετε δίκιο. Να περάσουμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Τελική ψηφοφορία. And it's closed. And it is widely... Μάλιστα, λοιπόν, ε, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται συγχαρητήρια στον συγκεκριμένο. are now waiting to proceed to the next item, which is the petition. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ο αναφέρον ε, θα καταφτάσει σε λίγο. Κάντε λοιπόν ένα μικρό διαλυματάκι, δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ. Now, I'm happy to welcome Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον αναφέροντα εδώ στην αίθουσα, Αντώνια Μπατάγλια, εξ ονόματος της Peace Link, που ε- την, για την αναφορά 7 του Οπότε ευχαριστώ να σας δώσω ευθύς αμέσω το λόγο και επίσης θα περιμένουμε κάποια στιγμή θα έρθει η μόνιμη αντιπροσωπεία ε, της ε, Ιταλίας ε, άλλοι γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν την ε, υπόθεση παρακαλώ ενημερώστε μας αλλά όχι παραπάνω από 5 λεπτά Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να σας μιλήσω για την Ήλβα, αυτή είναι την Χαλιβουργία, η οποία βρίσκεται στην πόλη στην Ιταλία και η οποία ήδη έχει καταγγελθεί για την ε, διαδικασία υπαραβάσης στην Επιτροπή. Πέρασε ένα μισό από τότε που ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στο Τάραντο, στον Τάραντο. Δηλαδή και εδώ πέρα έχουν περάσει κάποιοι μήνες και γίναμε μάρτυρες του ότι η κατάσταση δεν βελτιώθηκε καθόλου για να το πούμε και διπλωματικά. Και έχουμε ε, διάφορες δικαστικές ενέργειες έχουν γίνει και η Χαλιβουργία έχει μπει υπό κυβερνητική εποπτεία ε, βάσει του νόμου για το περιβάλλον, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το ότι θα συνεχιστεί η παραγωγή όσο γίνεται περισσότερο. Και έχουμε ένα νέο νόμο, ο οποίος είναι ακόμα πιο κακός για τον πληθυσμό, γιατί η διαδικασία Τις λειτουργία είναι εγγυημένοι, όμως έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι. Και επίσης ε, δεν ε, εφαρμόζονται αυτά που προβλέπει η υπερβολοντική άδεια. Η Ιταλική κυβέρνηση δεν ε, συμμορφώνεται με το κοινωτικό δίκαιο του Ιταλικού δίκαιο γιατί εγκρίνει κάποια νομοθετικά διατάγματα τα οποία είναι εις βάρος του πληθυσμού του Τάραντο γιατί κατοχυρώνεται έτσι το δικαίωμα στη δουλειά αλλά όχι στη ζωή και στο να μπορεί κανείς να αναπνεύσει. Επομένω, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ενισχυτική παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Γιατί τώρα έχουμε κάποιε υψηκαμίνε που έχουν κλείσει, αλλά αυτό δεν σταματά τη ρήπανση τη ατμόσφαιρας που προέρχεται από αλλού, από άλλε πηγέ. Και επομένω κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη σύμφωνα με ε, τις, ε, τους σωλήνες εκπομπής των καυσαρίων του εργοστασίου. Οπότε οι κάτοικοι εκεί και κυρίως τα παιδιά έχουν αφαιρεί στην τύχη τους ε, λόγω των εκπομπών του μολύβδου, της διοξίνης και άλλων βλαπτικών στοιχείων. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει ασθένειες αλλά και θανάτους. Επίσης, στη βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με οδηγία και το μητρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε εκπομπές από μόλιβδο, από κοβάλτιο, από διάφορες άλλες επικίνδυνες ουσίες και επομένως τώρα θα πρέπει να ληφθούν επιγόντως μέτρα και η θνησιμότητα είναι πάρα πολύ ψηλή κυρίως για τους ανηλίκους αλλά επίσης οι ασθένειες, αναπνευστικές ασθένειες ε, καρδιογγειακές ε, παθήσεις, γυναικολογικές, καρκίνη, όλα αυτά στον τάραντο τώρα ε, είναι πάρα πολύ αυξημένα και αυτό αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μα τι άλλο περιμένουμε, ποια είναι η λύση. Τι θα θέλουν να αλλάξουν το μέλλον της πόλης, τι θα γίνει άμα πεθάνουν όλα τα παιδιά. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική τραγωδία. Ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή. Έχουμε τη διαδικασία παραβάσει, αλλά αν δεν γίνει τίποτα θα επεκταθεί αυτή η κατάσταση και σε άλλες πόλεις και περιοχές. Καθυστερεί τις διαδικασίες η Ιταλία. και καθυστερούν την παροχή πληροφοριών και θέλουν να συνεχιστεί η παραγωγή από τη χαλιβουργία. Ενώ τα πράγματα χειροτερεύουν κάθε μέρα. Όμως συνεχίζουν και οι οικονομικές ζημίες στην βιομηχανία. Το δε μέλλον της Σίλβα είναι προβληματικό. Όμως την ύφη την πληρώνουν οι άνθρωποι με τη ζωή τους. Μάντρε Γκράτσια λέγεται εκεί η περιοχή αλλά αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι μόνο να ελπίζουμε ε, να τηρήσει η διεθνής κοινότητα τις δεσμεύσεις της να βοηθήσει τον Τάραντα. Η έγκριση λειτουργίας εκδόθηκε αλλά ποτέ δεν έγινε σεβαστή. Έχουμε ένα σωρό νομοθετικά διατάγματα τα οποία ουσιαστικά είναι εγγυήσει προς τη βιομηχανία για να συνεχίσει τη λειτουργία. Έχουν περιθωριοποιήσει τη δικαιοσύνη. Αυτό το που χρειάζεται είναι να κλείσει ένα σφαγιστή το εργοστάσιο και η Ιταλία δεν προτίθεται να κάνει τίποτα, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί το μέλλον του τόπου, εκεί, του Τάραντα. Και έχουμε πάρα πολλούς φορείς που ζητούν και απαιτούν κάτι να γίνει. Εδώ και χρόνια αυτό. Η κατάσταση της υγείας του κόσμου εκεί είναι πάρα πολύ ενισχυτική. Έχουμε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα ε, στην Ίσπρα, έχουμε ε, βίντεο, φωτογραφίες, όλη την τεκμηρίωση που απαιτείται. Δεν γίνεται τίποτα όμως. Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τις Ιταλικές αρχές να σταματήσουν ε, αυτήν την επικίνδυνη βιομηχανική δραστηριότητα και να έχει την υψίστη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δώσει ομένως όλα αυτά τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον, αλλά τελευταία φορά πιονίσαμε τον Οκτώβριο του 2014 με την Επιτροπή. Πέρασαν 7 μήνες. Από τότε είχαμε την αιτιολογημένη γνώμη, αλλά η κατάσταση συνεχίζεται, χειροτερεύει συνέχεια. Αυτό το οποίο σήμερα ζητούμε είναι να μας βοηθήσετε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί και να εξασφαλίσει ότι ό,τι χρειάζεται θα γίνει. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ καλή περιγραφή αλλά και για το γεγονός ότι τηρήσατε το χρονικό όριο, το οποίο συνήθω δεν συμβαίνει, σα διαβεβαιώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ιταλική μόνιμη προσωπία, όμως δεν κατάφερα να βρεθούν μαζί μας, γιατί πριν λίγο υπήρχε ένα ατύχημα. Αυτοκινητικό. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κ. Μαγκανάρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Όπως υπενθύμησε η εκπρόσωπος των αναφερομένων, η λειτουργία αυτής της χαλιβουργίας έχει αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής. Οκτώβριο του 2014 στείλαμε την αιτιολογημένη γνώμη στις ε, Ιταλικές αρχές, αλλά δεν απάντησαν τότε, απάντησαν τον Ιανουάριο του 2015 και στη συνέχεια είχαμε δύο συναντήσεις σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Συναντήσαμε στις Ιταλικές αρχές τον Μάρτιο του 2015. Μετά την τεχνική συνάντηση, οι υπηρεσίες μας ζήτησαν από τις Ιταλικές αρχές να στείλουν περαιτέρω έγγραφα. Γιατί ακόμα κάποια ζητήματα χρειάζονται διασάφηση από πλευράς των τελικών αρχών. Η τελευταία επικοινωνία έγινε στις 24 Απριλίου και η υπηρεσία μας αξιολογεί τώρα όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία μας διαβιβάζουν οι αναφέροντες. Όλα αυτά τα έγγραφα μελετώνται στα πλαίσια της ε, διαδικασίας επί η οποία και είναι η εξελίξη. Και όταν τελειώσει η αξιολόγηση από τη βάση αυτής της τεκμηρίωσης θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα πάντα στα πλαίσια της διαδικασίας επί Και σας ευχαριστώ. I thank you very much and now I open the for Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. κυρία Όκεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε αυτή την υπόθεση για αυτό το εργοστάσιο. Θυμάμαι πολλές ε, συνεδριάσεις και όταν Γιάννη ήταν τότε επίτροπος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά από περιβαλλοντικό ζήτημα ουσιαστικά περάσαμε κατευθείαν ε, στην αναγκαιότητα της ε, παραγωγής χάλιβα. Το θυμάμαι ως μια πολύ κακή εμπειρία. Όμως δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι έγινε με λεπτομέρειες. Όμως έχουμε την εντύπωση ότι ο Επίτροπος Ταγιάννη ερχόταν εδώ, πήγαινε στην Ήτρε, τα έφερε όλα πάνω κάτω. υπήρχε υποτίθεται και μία νομοθετική πράξη. Μετά η Ιταλική κυβέρνηση άλλαξε τους νόμους τους ώστε να καταστεί νόμιμη αυτή η διαδικασία. Μπορεί και όμως και η χαλιβουργία να γίνει με αξιοπρεπή τρόπο. Αντί να επιμένουμε σε αυτό, τώρα η Επιτροπή, τώρα δεν είναι πλέον ο Ταγιάννη, ευτυχώς, είναι ένα μέλος που του δίνει μόνο μια ψήφο κάπου. Όμως και πάλι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει με δίκαιο τρόπο τις αναφορές αυτές. Έχει έρθει πραγματικά η ώρα να αντιδράσουμε σε αυτές τις αναφορές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαχτά έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την ε, αναφέρουσα. Χαίρομαι που ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, γιατί και εγώ πήγα στον Τάρατα πέρυσι τον ε, Δεκέμβριο. Έχω και μία ε, νομοδότηση πρωτοβουλία για τις μεθόδους βασικής παραγωγής που θα παρουσιάσω σύντομα και επισκέφθηκα την περιοχή και συνομίλησα με κατοίκους της περιοχής που είναι θύματα πολύ σημαντικών ασθενειών. Μάλιστα υπήρξαν και πολλοί θάνατοι. Και υπάρχουν και κάτοικοι, ένα τμήμα του πληθυσμού που υπό το πρόσχημα ε, του εκβιασμού σε ό,τι αφορά την απασχόληση λέμε ότι μπορούμε να κλείσουμε το εργοστάσιο γιατί θα χαθούν θέσει εργασία. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέσει και να πω είναι το ένα ή το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο είναι δυνατά. Η κατάσταση στην περιοχή αυτή, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι η οικογένεια Ρίβα ε, δεν έχει τηρήσει ούτε περιβαλλοντικούς νόμους, ούτε κανένα άλλο νόμο. Κατάλαβα λοιπόν ότι το Ιταλικό κράτος είχε δεσμευθεί να επενδύσει περίπου 2 δις ευρώ για να επιστρέψει το εργοστάσιο, να τεθεί και να τηρήσει ε, τα πρότυπα τα περιβαλλοντικά. Από ό,τι βλέπω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η παραγωγή είναι 60% αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να ρηπαίνει το περιβάλλον. Θα ήθελα πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προσφύγει εναντίον του Ιταλικού κράτους, να δούμε τι συμβαίνει με αυτές τις απαραίτητες επενδύσεις και να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των ε, επενδύσεων. Γιατί πραγματικά δεν είναι διαπραγματεύσιμη υπερβολική ε, διάσταση, όμως πρέπει να σταματήσει και αυτός ο εκβιασμός ότι φορά την απασχόληση. Δεν είναι το ένα ή το άλλο, είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Θα μπορούσα να απαντήσω, όχι ακόμα. Πιο μετά. Θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Κύριο. Ευχαριστώ. Είμαι Ιταλός Ευρωβουλευτής και θεωρώ ότι Βεβαίω και είναι αδιαπραγμάτευτη η δημοσία υγεία. Φυσικά και η ζωή είναι πάνω απ' όλα και πάνω από το δικαίωμα στη δουλειά. Μα είναι δυνατόν να αμαυρώνεται ε, έτσι η εικόνα της ε, χώρας. Ε, εγώ ανήκω στον πολιτικό συνασπισμό που αστηρίζει την κυβέρνηση, οπότε είμαι υπέρ των θεσμών, των θεσμών οργάνων της χώρας, Οπότε βλέπουμε πώ έχει η κατάσταση στον Τάραντο, τι γίνεται με την Ήλβα, κάθε μέρα πεθαίνει ο κόσμο, κάθε μέρα αρρωσταίνει ο κόσμο και κάθε μέρα δεν δίνει δεκάρα η Ιταλική κυβέρνηση για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ούτε ενδιαφέρεται και η περιφερειακή κυβέρνηση και όλα συνεχίζονται σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Έτσι λένε, αλλά ίσω δεν είναι έτσι, γιατί θα πρέπει βέβαια να δούμε το ότι Φυσικά και πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή, πάνω απ' όλα είναι, πάνω απ' όλα τα συμφέροντα και συμφωνούμε από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να δεχτώ εδώ πέρα σε την αίθουσα να λέγεται ότι, ότι ασκεί πιέσει στη δικαιοσύνη η κυβέρνηση για να μην κλείσει το εργοστάσιο. Μα αυτές οι διατυπώσει είναι πάρα πολύ έντονε και απόλυτε. Μα ε, άλλο, άλλο η δικαιοσύνη και άλλο η κυβέρνηση. Εγώ Θέλω να υπερασπιστώ του Ιταλικούς θεσμούς. Και έχουμε και την ε, περιφέρεια που έχει αρμοδιότητες και για την ε, δημοσία υγεία και πολλές φορές είναι αλήθεια ότι οι υπηρεσίες κινούνται πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε. Και αυτό το οποίο σίγουρα επιβάλλεται είναι τα θεσμικά όργανα να κάνουν ό,τι πρέπει. Όπως και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι' αυτό και νομίζω θα πρέπει να μην ανοιχτή αναφορά και θα πρέπει επομένως να κινηθεί η κυβέρνηση με ταχύτερους ρυθμούς. Όμως δεν είναι δυνατόν εδώ να μαυρώνεται ε, έτσι η εικόνα της χώρας και να λένε ότι κάθεται και παρακολουθεί αμέριμνη η κυβέρνηση το να πεθαίνει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πρόεδρος. Επομένη. Κυρία Εύη. Εγώ θα ήθελα να σας τονίσω ότι φταίει και η κυβέρνηση. Μα είναι φανερό. Αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο. Καταστρέφεται και η περιοχή και αυτό έχει κρατήσει τόσο καιρό. Και ουδέποτε έχουν κάνει οτιδήποτε για να αλλάξει η κατάσταση. Φερμπίν, αυτό το οποίο δεν έχει γίνει είναι να γίνει μια επιδημιολογική ανάλυση των εκπομπών και να δούμε πώς όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί δρούν σωρευτικά και όχι μόνο ξεχωριστά κάθε μία της ουσίας όπως αναφέρθηκε. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει μόνο ένα κομμάτι της εικόνας και του σκηνικού. Άρα έτσι αυτό να δούμε τι γίνεται για το σύνολο των εκπομπών της Χαλιβουργίας. τι γίνεται, πόσο παραβλάπτεται το έδαφος, ε, αυτή η διοξίνη που καταλήγει στα γεωργικά προϊόντα, στα είδη διατροφής, ό,τι τρώει ο κόσμος. Υπάρχει η ρήπανση της ατμόσφαιρας, αλλά και του εδάφους. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία όντως έχουν αναφερθεί, αλλά όχι σοβαρά. Έχουμε επίσης το τελευταίο νομοθετικό διάταγμα υπαριθμό 7, δυνάμει του οποίου δεν δικαιούνται οι φυγέντε αποζημίωση. Τα ξέρει εδώ η παρακαθήμενη στις λεπτομερίες του τα ζητήματα. Μιλάμε για 30 εκατομμύρια τα οποία έχει αξιώσει η πολιτική αγωγή. Πρόκειται για τις οικογένειες όσων πέθαναν. Και μιλούμε για χιλιάδες κόσμου. Επομένως, ας αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ασκήσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πίεση, μπάσκετ και αλλάξει τίποτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την αναφέρουσα που ήρθε εδώ για να μας περιγράψει αυτή τη δραματική κατάσταση που αφορά την πόλη μου. Γιατί και εγώ από τον Τάραντα έρχομαι. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από την κυβέρνηση και έχουν αποφύγει να λάβουν κάποιες ε, αποφάσεις πάρα πολύ κρίσιμες που έχουν σχέση με το περιβάλλον αλλά και την ε, υγεία μιλάμε ε, ότι η ιστορία ξεκίνησε το 2011. Οι δικαστικές αρχές ε, επελύσαν το 2012. Πάρα πολύ λίγα έγινε τόσο ώστε να φροντίσουν τον κόσμο, να φροντίσουν το περιβάλλον, να προστατεύσουν τελικά και άλλες οικονομικές δραστηριότητε. Ε, και γι' αυτό η κυβέρνηση τελικά κατέληξε σε κάποια νομοθετικά διατάγματα. Φρενάρισε τη δικαιοσύνη. Τελικά δεν έκαναν τίποτα. Και έχουμε επιδημιολογική μελέτη ε, όπως είπε η συνάδελφος, και μιλάμε για 13 χρόνια. Ε, μιλάμε για 13 ε, χρόνια και έχουμε 30 νεκρούς κάθε χρόνο. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαριστεί περισσότερο το θέμα πόσο ρηπαίνεται η ατμόσφαιρα από τη χαλιβουργία. Και γι' αυτό και έχουμε εκφυλιστικά φαινόμενα που υφίσταται ο πληθυσμός. Αρρώστιες και θανάτους. Εάν αυτό δεν λέγεται ε, περιβαλλοντικό ε, δυστύχημα, περιβαλλοντική τραγωδία τι να είναι και οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα σταματήσει αυτή η υπόθεση και θα πρέπει επομένω την επόμενη τριετία να μην συνεχιστεί η δραστηριότητα της χαριβουργίας. Αυτά τα έχουμε πει και έχουμε και κάποια αίτηση γι' αυτό από τον φορέα των ε, γιατρών για το περιβάλλον. Έχουμε επομένω ε, καρκίνους διαφόρων μορφών, έχει ε, αυξηθεί η θνησιμότητα και έχουμε ένα σώρο λοιπόν ε, ε, όγκους που βγαίνουν στο, στον κόσμο και επίσης η διατροφική αλυσίδα έχει ε, και ακόμα και τα, και τα έμβρια επίσης υφίστανται ε, βλάβες στην υγεία τους. Και βέβαια κάνουν ή τις κυβέρνησες ότι αναλαμβάνουν ενέργειες, αλλά δεν είναι αλήθεια. Έχουμε ακόμα και απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που κήρυξε αντισυνταγματικό το πρώτο νομοθετικό διάταγμα που αφορά την Ήλβα. Δεν έχουν αφήσει την υπηρεσία υγείας να επιληφθεί. Πρόκειται επομένω για μια τραγωδία που αφορά την υγεία, αφορά το περιβάλλον και επομένως σύμφωνα με εκτιμήσεις έχουμε ένα σωρό όγκους που αναπτύσσονται μόνο, ε, μόνο με το να αυτόν τον αέρα. Και ε, έχουμε 22.000 κόσμου που ζουν γύρω και έχουν υποστεί βλάβες οι 12.000. Τώρα, Ποια είναι τα αιτήματά μας. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επιληφθεί γιατί είναι προβληματική ε, αυτή η βιομηχανία και μιλάμε τώρα για ζημίες ενός δισεκατομμυρίου και έχουμε την οδηγία 75 του 2010 ε, ούτως ώστε να κλείσουν ε, οι βιομηχανίες που μολύνουν. Είναι bad company αυτή η εταιρεία. Έχουμε και την οδηγία 35 του 2004. Επομένως κάποιος θα πρέπει να σταματήσει αυτή την κατάσταση και να μην φροντίζει κάποιος αυτή την εταιρεία και να την αφήνει να λειτουργεί όπως κάνει η κυβέρνησή μας. Είπαμε ότι θα πρέπει να διατεθούν 120 εκατομμύρια ε, ούτως ώστε να υπάρξει κάποιος αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνει η ταλική αντιπροσωπεία, θα πρέπει ε, κατά αυτόν τον τρόπο να σταματήσει η διασπάθηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ε, αυτό ισχύει γενικά, αλλά ακόμη περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση του Τάρεντα. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να κρατήσει κανείς το χρονικό όριο όταν έχει τόσο μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, την οποία και προφανώς έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή και τώρα το λόγο έχει ο κ. Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα η οποία πραγματικά έχει θέσει αυτό το σοβαρότατο ζήτημα στην Επιτροπή μας. Διότι πρόκειται για ένα θέμα που όπως αναλύθηκε και κυρίως από τις ε, συναδέλφους ε, από την Ιταλία ε, μιας περιβαλλοντικής τραγωδίας όταν έχουμε τη λειτουργία αυτής της βιομηχανίας η οποία όχι μόνο ρηπαίνει το περιβάλλον αλλά είναι πλέον επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Έχουμε μόλυνση του αέρα και του εδάφους. Επομένως πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά να υπάρχει προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσει να συμβαίνει αυτή η τεράστια περιβαλλοντική τραγωδία. Το δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την ε, αναφορά είναι η αξιοποίηση από διάφορες επιχειρήσεις και κυρίως από τη συγκεκριμένη Χαλιβουργία ε, του προβλήματος απασχόλησης που υπάρχει σε διάφορες περιοχές όπου πιεζόνται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και απειλούνται ότι αν κλείσει μια δραστηριότητα ή μια βιομηχανική δραστηριότητα ε, θα μείνουν χωρίς δουλειά. Επομένως πιέζουν τους ίδιους τους εργαζόμενους να απαιτούν να λειτουργούν βιομηχανίες και εκμεταλλεύσεις οι οποίες μπορεί να παραβιάζουν την ομοθεσία του περιβάλλοντος αλλά οι ίδιοι αγωνιούν για τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει αντίθεση, πιστεύω, μεταξύ της δημόσιας υγείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της απασχόλησης. Εάν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να έχουμε περιβαλλοντική προστασία και απασχόληση. Το τρίτο θέμα που τίθεται είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν πλέον έτσι οι χαλιβουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γίνει επένδυση σε όλες τις χαλιβουργίες, διότι αυτή τη στιγμή κλείνουν χαλιβουργίες στην Ελλάδα έχουμε πάρα πάρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι είναι, ε, έχουν βρεθεί στην ανεργία, άλλοι υποαπασχολούνται και πρέπει να έχουμε πραγματικά ένα αναπτυξιακό σχέδιο για λειτουργία χαλιβουργία στην Ευρώπη, η οποία όμως θα σέβεται τους όρους τους περιβαλλοντικούς. Αυτή είναι η νέα κατεύθυνση την οποία πρέπει να δούμε. Επομένως αυτό είναι ένα τρίτο συμπέρασμα που βγάζουμε από αυτή την αναφορά. Η πρότασή μας είναι ότι αυτή η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή, πρέπει να πιεστούν οι Ιταλικές αρχές για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πρέπει φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. And now the floor... Και τώρα το λόγο έχει η Μάγκρετ Άουγκεν, αλλά για λίγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε κατευθείαν στο δικαστήριο για κυρώσει πλέον. Γιατί το έχουμε το θέμα αυτό τόσο πολύ καιρό. Και τώρα να καλέσουμε και πάλι τη μηχανία να ανταποκρινθεί στου κανόνες. Είναι σαν να λέμε να μην κάνουμε τίποτα. Τώρα θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Έχουμε τόσε πολλές παραβάσει εδώ. Επιτέλου θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθημα, ένα αίσθημα κατεπήγοντος. το όλο θέμα, το όλο σύστημα διακυβέρνησης στην Ιταλία είναι αδιαφανές. Αυτό αντιμετωπίζουμε και εδώ τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοζολίνο. Θα πρέπει να δούμε και να αποφασίσουμε τι θα γίνει σε σχέση με αυτό το οποίο εκκρεμεί τόσους μήνες. Έχουμε εδώ πέρα όλη αυτή την τεκμηρίωση από το 2013-2014 Άρα να δούμε τελικά πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία η παραβάση. Να αναπευθεί τελικά στην Επιτροπή ε, ο φάκελος και να δούμε κάπου θα καταλήξουμε αφού εμπλακούν όλοι οι τα θεσμικά όργανα. Έχουμε τώρα το, το πρόβλημα αυτό το οποίο αφορά γενικότερα τη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Ευθύνες έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Εθνική Κυβέρνηση αλλά και ο ιδιωτικό τομέα γιατί ξεκίνησε κρατικό αυτό το εργοστάσιο. Κατόπιν η Χελβοργία έγινε ιδιωτική, επομένω είναι περίπλοκη ε, η διαδικασία και το, μάλλον το νομικό καθεστώ τη ε, διαχείριση τη ε, Χαλιβουργία. Οπότε βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το θέμα είναι το πώς τον έχουμε αυτού του είδους τα προγράμματα αποκατάστασης. Αλλά εδώ πέρα μιλούμε για βιομηχανία πάρα πολύ μεγάλη. Και βέβαια για να γίνει αποκατάσταση πρέπει να υπάρξει διακοπή λειτουργίας. Και τι θα γίνει με όλες τις χιλιάδες των εργαζομένων. Αν μιλάμε εδώ πέρα για 14-15 χιλιάδες εργαζομένους. Επομένως το θέμα είναι πολύ πολύ περίπλοκο. Άρα, βεβαίω και θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ πέρα ε, χρεοκόπησε ως προς το πρόβλημα η κυβέρνηση και η πολιτική. Αλλά αυτό όμως τελικά είναι θέμα όλης της Ευρώπης. Να, αν δείξει κανείς τόλμη, τι θα πρέπει να πει. Πάντως, πρόκειται για δύσκολη κατάσταση. Και δύσκολη θα είναι και η λύση. Και δεν αρκεί αυτή η διαδικασία επί παραβάση. Ας πούμε, αποφασίζεται αύριο να κλείσει η χαλιβουργία. Όμως, έχουμε τις μελέτες τις ε, επιδημιολογικές, έχουμε το θέμα της αποκατάστασης, αλλά είναι λύση αυτό. Επομένως, τι θα έλεγα εγώ. Θα πρέπει να κάνουμε τα ζυγίσουμε. Θα πρέπει να αναπαιμφθεί η υπόθεση στην Επιτροπή Αναφορών όταν τελειώσει ο διάλογος ο θεσμικός για να δούμε σε ποια φάση θα έχει φτάσει η διαδικασία της, ε, της παράβασης. Είπαμε ότι ακόμα δεν έχει επιτροπή αρκετά στοιχεία. Ούτως ώστε. Τελικά, πέραν των καταθέσεων και μαρτυριών που έχουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι αποφάσεις μπορούν να πάρουν τα θεσμικά όργανα. Ό,τι και να πει κανείς, θεμητό είναι. Κάθε αξιολογική κρίση είναι θεμητή. Όλα αυτά είναι λογικά. Αλλά τελικά η συζήτηση δεν καταλήγει πουθενά. Και το σούτο μάλλον είναι σοβαρό αυτό, μια που το πρόβλημα είναι τόσο τόσο σοβαρό. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στην αναφέρουσα. Παρακαλώ. Και Καταλαβαίνετε ότι εδώ η Επιτροπή μας ε, δείχνει σημαντική κατανόηση για αυτή την υπόθεση, γιατί είναι η Ευρώπη και όλοι νοιαζόμαστε για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω καταρχήν όσον αφορά αυτά τα στοιχεία. Αυτό που είπατε για τα δύο δις, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Προβλέπει το τελευταίο νομοθετικό διάταγμα σχετικά. 400 εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί. Και με έχουμε τα 1,8 δις που αποφασίστηκαν ούτως ώστε να έχουμε την αποκατάσταση του Τάραντα. Όμως αυτά δεν είναι επαρκή και πάντως θα πρέπει τον κύριο Ντεμό τον ευχαριστήσω και θα πρέπει να πω στον κύριο Κοτσολίνο κάτι όσον αφορά το θέμα των ευθυνών ε, και την χρεοκοπία της πολιτικής γιατί θυμάμαι ότι στην πόλη ήμασταν βέβαιοι ότι η θνησιμότητα ήταν τόσο τόσο υψηλή και συνέχεια αυξανόταν η θνησιμότητα των ανηλίκων και αυτό ήταν αναποτελεσματικότητα των αρχών που δεν μπορούσαν κάτι να κάνουν για την Ήλβα. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαλιβουργία. Ναι, είναι τεράστια η πρόκληση του να έχουμε αποκατάσταση τόσο μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι όμως προφάσεις και δικαιολογίες. Αλλά το θέμα είναι ότι η ζωή των Ιταλών θα έπρεπε να έχει την κύρια προτεραιότητα για πάσα ανάληψη δράσης. Καλά. Η διαχείριση της χαλιβουργίας, της Σίλβα, ήταν παράξενη τα τελευταία χρόνια. Αλλά αν δεν μπορεί να κάνει τη διαχείριση το κράτος, ποιος θα την κάνει, γιατί υπάρχουν θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και οι επιπτώσεις τώρα είναι τέτοιες που είναι αφόρητες. Οπότε τελικά θα πρέπει κανείς να αποφασίσει ή θα τακτοποιήσει την κατάσταση, κάτι το οποίο θα χρειαστεί χρόνο ή από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε το ότι την ύφη την πληρώνει ο πληθυσμός για να έχει αυτή την παραγωγή η Ιταλία. Γιατί έχουμε τους ανηλίκους που έχουν αυτή την σημότητα και τελικά το ίχνος, το αποτύπωμα αυτής της ε, διοξίνης πάει σε όλη την Ιταλία και αυτό ε, δεν είναι αξιολόγηση, δεν είναι γνώμη. Υπάρχουν μελέτες ότι το, το αποτύπωμα αυτό ε, της διοξίνης έχει φτάσει μέχρι το Μιλάνο και έχουμε την επιδημιολογία, έχουμε επιστήμονες που μας δίνουν τα στοιχεία. και η ζημιά στην υγεία των κατοίκων του Τάραντα δεν αφορά μόνο τους σημερινούς κατοίκους. Είναι κάτι που θα αφορά και το μέλλον. Άρα, είπαμε ότι έχουμε υποβάλει φωτογραφίες και βίντεο από ένα μαύρο σύννεφο που κρέμεται πάνω από την πόλη και ορίζεται εκεί. Επομένως θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Είδατε, είπαμε, πληρώνουν την ύφη κάτοικοι του Τάραντα. Ευχαριστώ κύριε Μάτο. Η κατάσταση όμως είναι απαράδεκτη. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Εφόσον ακόμα υπάρχει εκπρόσωπος ε, της Κομισιόν και είναι ενδιαφέρον το ζήτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να επανέλθετε. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να δώσω για πολύ λίγο στην κυρία Νταμάτο. Όμως τώρα που ακούσατε και τους συναδέλφους, καλό θα ήταν αν μπορείτε κι εσείς ε, να συνοψίσετε, αλλά και να πείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Ποιε είναι οι προθέσει σα. Η κυρία Νταμάτο πρώτα. Χρειάζεται υπευθυνότητα, χρειάζεται θάρρος. Μιλάμε για την υγεία και μιλάμε και για την οικονομία. Μιλάμε για 14.000 εργαζόμενους, μια ολόκληρη πόλη είναι η γεωργία, είναι ο τουρισμός. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πεθαίνουν. Έχουμε 100.000 κατοίκους στην πόλη οι οποίοι υφίστανται όλα αυτά. Έχουμε 43% ανεργία. Άρα τι γίνεται με την υγεία. Πού είναι η οικονομική ευημερία που μας δίνει αυτή η μεγάλη εταιρεία. Έτσι είναι η κατάσταση. Θα πρέπει να κλείσει η επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να παράγει το χάλιβα στον Ταρόντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Μαχτά. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα. Εφόσον μιλάμε για ευθύνε και τι αδυναμίε τη Ευρώπη, υπάρχει και μία στο δικαστικό επίπεδο, γιατί ε, η Ρίβα έχει βρει καταφύγιο στην Αγγλία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την, ε, τις δημόσιες αρχές και τις ευθύνες της, αλλά πρώτη ευθύνη και πρώτος υπεύθυνος είναι η ίδια επιχείρηση. Και επαναλαμβάνω και ευχαριστώ και τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένω ότι η επόμενη έκθεση που θα παρουσιαστεί αφορά ακριβώ αυτό το ζήτημα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την μέθοδο λειτουργία μα. Και δεν πρόκειται μόνο για μια χαλιβουργία που δίνει απασχόληση ε, σε βάρο ε, τη ανθρώπινη ζωή ή του περιβάλλοντος, είναι και τα δύο. Ελπίζουμε να ακολουθηθεί ο προσανατολισμός που θα προτείνουμε σε επόμενες εβδομάδες. Ναι, κάτι μόνο. Το... Α, η Πρόεδρος, συγγνώμη, αλλά δεν έχετε το λόγο. Είναι μια πολύ σπάνια κατάσταση. Δεν έχουμε περιορισμό στον χρόνο. Έχουν ζητήσει δύο συνάδελφοι ε, ακόμα το λόγο και να φερολογήσουν ο κύριος Κοζολίνο και ο κύριος Μαριάς. Για ένα λεπτό καθένας και μετά θα θέσουμε τέλος στον κατάλογο μελετών. Νομίζω ότι έχουμε πει όλα. Κυρία Πρόεδρε, <clears throat> νομίζω ότι εδώ αναδεικνύεται η αντίφαση ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της απασχόλησης. Αλλά στην πράξη δεν μπορεί να υπάρχει αντίφαση. Δεν μπορεί να έχουμε λειτουργία βιομηχανίας που καταστρέφει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα έθεσαν οι συνάδελφοι ένα θέμα. Τι θα γίνει με τους 14.000 εργαζόμενους. Θα μείνουν άνεργοι. Άρα λοιπόν το θέμα είναι συγκεκριμένο. Πρώτον, άμεσα μέτρα για την τήρηση της νομοθεσίας και δεύτερο, όπως είπε ο συνάδελφος, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης της χαλιβουργίας στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε τον κύριο Ντράγκη που δίνει 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ για αγορές ομολόγων και να μην έχουμε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν στη βιομηχανία και όχι να έχουμε μια οικονομία καζίνο με αγορές απλά ομολόγων. Άρα λοιπόν συμπέρασμα και νομίζω αυτό πρέπει να το στείλουμε και στην Επιτροπή την Ίκον και σε άλλες επιτροπές. Πρέπει να επενδυθούν άμεσα κεφάλαια για βιομηχανία για τη χαλιβουργία η οποία όμως θα σέβεται το περιβάλλον. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα γιατί έχουμε τέτοια προβλήματα όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που κλείνουν οι βιομηχανίες μένουν άνεργοι τόσοι άνθρωποι ενώ υπάρχουν κεφάλαια και πρέπει να επενδυθούν. Αυτό είναι το βασικό. Αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εδώ και τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Now the floor goes. Το ναι, επιμένω όμως ε, στο εξή. Δεν θέλω να μπω στην ουσία τη συζήτηση. όμως εδώ, στην κουβέντα που κάνουμε σήμερα, να πω τη γνώμη μου. Ίσως μπορούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις ε, και πιο αποφασιστικά μέτρα δεν πρόκειται να αμφισβητήσω τα στοιχεία που ακούσαμε σε ό,τι φορά την δημόσια υγεία στο Τάραντο ή τις γενικότερες επιπτώσεις. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αν δεν θέλουμε αυτή η αναφορά ε, να μείνει μόνο στο γράμμα και να μην μπει στην ουσία, θα ήθελα, Πρόεδρε, να ζητήσω να επιστρέψει η Επιτροπή και να επανεξετάσει ε, αυτή την αναφορά. Εάν υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη παραβάση, να δούμε τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε. Για να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ε, να δεσμευτεί και να επιληφθεί της κατάστασης. Αυτή τη χρονική στιγμή ξέρουμε ποιε είναι οι απόψει, υπάρχει διαφορά απόψεων και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα σε διαφορά του πόρου. Δεν έχουμε του πόρου να ε, ενεργήσουμε βάσει ενό καθαρότερου προγράμματο. Δύο δι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ τη χώρας, σε οικονομικούς όρους δηλαδή, θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης πόρων. Σε ό,τι αφορά και την ε, κερδοφορία και τη βιωσιμότητα και των επενδυτών. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Δεν πρέπει όμως να χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται με αυτή την υπόθεση να επιστρέψουμε σε μία συζήτηση με την Επιτροπή και την κυβέρνηση για να έχουμε καλύτερες λύσεις. Ε, εντάξει, ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσατε τους συναδέλφους, ακούσατε τις προτάσεις ε, που έθεσαν Τώρα, αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω τι γίνεται. Να σας ε, πω τι περιέχει η ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ιταλικές Αρχές. Αξιολογούμε το τελευταίο έγγραφο που λάβαμε στις 24 Απριλίου και θα αξιολογήσουμε και θα εκτιμήσουμε όλα αυτά τα οποία λάβαμε και από την αναφέρουσα. Μόλις γίνουν λοιπόν οι εκτιμήσεις αυτές ε, για το σύνολο των πληροφοριών θα ληφθεί η απόφαση. Το, τον Οκτώβριο του 2014, όπως σας είπα, ε, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και το βήμα είναι το να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά, όπως σας είπα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι αξιολογήσεις, οι εκτιμήσεις. Τώρα, στην προκειμένη φάση δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να κλείσω το θέμα αυτό, αν μου επιτρέπετε, με έναν τρόπο που θα μας ε, αποδειχθεί επικοδομητικός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εδώ επί σειρά ετών. Ο κόσμος υποφέρει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και η Επιτροπή μας λοιπόν θέλει κατεπηγόντως να διορθώσει την κατάσταση γιατί η δημόσια υγεία δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο. Το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Τι μας λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πριν από μία εβδομάδα λάβαν νέα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν αντιπρόσθετα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επανέλθει με τις πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα προθεσμία να τεθεί όμως πριν τα τέλη του Ιουνίου θα πρέπει να δοθεί πληροφορίε στην Επιτροπή μας για την υπόθεση αυτή. Γιατί τα λάβατε πρόσφατα τα στοιχεία και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει ακόμα σχετική ανάλυση. Αν όμω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να έλθει και πάλι στην Επιτροπή μα. Πότε. Σε δύο μήνε, σε δύο μήνε, έχετε δύο μήνε. Με μια πλήρη ανάλυση τη κατάσταση θα ήμασταν ικανοποιημένοι και θα μπορούσαμε να βρούμε τις περαιτέρα προτάσεις για τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Συμφωνείτε, συνάδελφοι? Πολύ ωραία. Εντάξει, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να, υπάρχει, να είναι μαζί μας σήμερα η Ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία, αλλά τι να κάνουμε. Στέλνουμε τις ε, ευχές μας ε, και τις καλύτερες ε, ευχές μας στο άτομο που είχε το ατύχημα αυτή σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. The next case that we Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, 21 του 2013 του Πιέρο Μπρούνι για την μόλυνση της ελίμνης Μολσένα. Αναφορά 21-91-2013. Καλώς ορίσατε κύριε Μπρούνι, είσαστε εκπρόσωπος του Λάκο την Μολσένα της Σχετικής Ένωσης. Σας δίνω το λόγο και σας ε, ζητώ σας παρακαλώ να κάνετε προσπάθεια να τηρήσετε το χρονικό όριο. 5 λεπτά έχει στη διάθεσή σας. Ε, Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκίνησε η διαδικασία παραβάση κατά της Ιταλίας γιατί δεν έχουν θεσπιστεί τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να προστατευτεί αλλά και να αποκατασταθεί η περιοχή της ε, ε Λίμνης Μπολσένα. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος και η διαδικασία επί παραβάση αφορά την περίοδο από το 2008. και προκαλείται ρήπανση στην λίμνη από τα λίμματα αλλά και από το αρσενικό το οποίο εκεί εκχύεται και είναι καρκινογόνο και αφορά και το δίκτυο του υδροδότησης για το πόσιμο νερό. Είναι ιδιόμορφη η κατάσταση στη λίμνη, γιατί είναι ηφαιστειακού τύπου και εκεί έχουμε μια επιφάνεια που αφορά την, τον υδροφόρο ορίζοντα. Και εκχύεται τελικά η λίμνη στον Στίβερη και κατόπιν στην θάλασσα. Έχουμε αυτή την μαύρη γραμμή που υιοθετεί αυτή την περιοχή και έχουμε υπόγεια ύδατα και επιφανειακά ύδατα τα οποία θίγονται και έχουμε το βρόχινο νερό Οπότε και στην διαδρομή του το νερό ε, περνάει από περιοχές όπου ε, μολύνονται από λιπάσματα, τα οποία που είναι γεμάτα φόσφορο. Έχουμε παραγωγή του αρσενικού, το οποίο επίσης μέσα των υπογείων υδάτων, αλλαγέ των επιφανειακών, ε, καταλήγει στην λίμνη και κατόπιν στη θάλασσα. για να προστατευτούν από τα λίμματα η ε, οι, οι, δήμοι εκεί γύρω υπάρχει Υπάρχουν κάποια αγωγή συλλογή λιμάτων. Βλέπετε που είναι. Αλλά εκεί έχουμε και σπίτια, έχουμε κάμπινγκ, εστιατόρια. Οπότε από εκεί έχουμε επίσης ε, φόσφορο και άλλα πλοκτικά υλικά τα οποία εξηγούνται στην λίμνη. Έχουμε επομένω ε, αυτόν τον αγώ συλλογής λιμάτων ο οποίος είναι σε πάρα πολύ κατάσταση και επί χιλιόμετρα εκτείνεται ε, γύρω γύρω στην ε, λίμνη και προκαλεί την υπερχείληση και θα πρέπει να δούμε τι μέτρα χρειάζονται και ο φόσφορος όλο ένα και αυξάνεται ήταν 8-9 μικρογραμμάρια ένα λίτρο πριν από λίγες μέρες μετρήθηκε και έφτασε στα 15 μικρογραμμάρια. Η κατακλείδη από το 2008 μέχρι σήμερα δεν γίνει καμία κίνηση βελτίωσης. Δεύτερον, τα μέτρα της ε, αποκατάστασης θα έπρεπε να μειώσουν τον ε, φόσφορο και να κατέβει η περιεκτικότητα κάτω από τα 10 μικρογραμμάρια ένα λίτρο. Αυτός ήταν ο στόχος. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με το αρσενικό. Δεξιά βλέπουμε το καρκινογόνο υλικό το οποίο προέρχεται από την λεκάνη του Τίβερη κάτω από την ε, λίμνη. Ανεβαίνει στην επιφάνεια ε, ζεσταίνεται και με το αυτό φαινόμενο και μετά κατεβαίνει ψυχρότερο. και επομένως λόγω του τύπου του εδάφους πολύ από αυτό το αρσενικό καταλήγει στην λεκάνη της λίμνης. Επομένως, είπαμε ότι ο στόχος είναι να καταλήξουμε στα 10 μικρογραμμάρια φωσφόρου ανά λίτρο. Επίσης, ενώ εδώ προβλέπεται να είναι πόσιμο το νερό της λίμνης, κάτω από τα 10 μικρογραμμάρια, με μιλήσει και κατόπιν. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το αρσενικό στη λίμνη, το οποίο ε, ε, και ακόμη και στα 6 μικρογραμμάρια ξαναμπαίνει στο πόσιμο νερό. Οπότε έχουμε τελικά θα πρέπει να διευθυνθεί η κατάσταση που είναι παράδειγμα και θα πρέπει επομένω να δούμε το, το πώ θα υπάρξει ενθάρρυνση για ε, βιολογικέ καλλιέργειες στην ε, Λίμνο Λεκάνη και εκεί στο Βιτέρμπο θα πρέπει να γίνει κάποια ευρωπαϊκή προσπάθεια οπότε θα πρέπει να πιστοποιηθεί από επίσημο οργανισμό το ότι όλα εκεί τα, τα σπίτια, ε, τα καταστήματα, ότι λειτουργούν, συμμορφούν με την νομοθεσία και δεν ε, εκχύουν λίμματα στην λίμνη. Οπότε ολοκληρώνοντας θα σου πω ότι κάτι πρέπει να γίνει και με την επιφάνεια αλλά και με το ε, βυθό της λίμνης. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάρε και λος Μαγκανάρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακριβώς όπως σας είπε ο αναφέρον, ήδη βρίσκεται να εξελίξει μια διαδικασία επί παραβάση για την ε, λίμνη. Και ουσιαστικά τώρα πρόκειται ότι είμαστε στη φάση της έρευνας για να καταλήξουμε τη διαδικασία επί παραβάση. θα ολοκληρωθεί τον ε, Απρίλιο. μόνο τον ε, Απρίλιο η έρευνα και είπαμε ότι στην λίμνη Μπολσέν έχουμε πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτα-πρώτα έχουμε το ότι ε, τα, τα λίμματα, τα αστικά δεν υφίστανται την δέωση επεξεργασία όπως είπε ο αναφέρον. Και επίσης έχουμε ρήπανση που προέρχεται από την γεωργική δραστηριότητα, από ε, τα, το, το φόσφορο από ό,τι περιέχουν τα λιπάσματα. Θα πρέπει κάτι να γίνει επομένως για να ανασχεθούν αυτές οι δύο πηγές της ρήπανσης που αποτελούν την περιβαλλοντική πίεση επί της λίμνης ε, γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να σωθεί η ποιότητα του νερού. Όπως προβλέπει ο ΙΕ 2060. Έχουμε επομένω τα αστικά λίμματα που καταλήγουν στη λίμνη και σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές οι εργασίε ε, για, τον εξυγχρονισμό του χώρου επεξεργασίας αυτών έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει πριν λίγο και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2017 αυτό τόσο εξυγχρονισμός τη μονάδα επεξεργασία των κλιμάτων. Θα παρακολουθούμε επομένως την πρόοδο των εργασιών και ίσω θα θυμάστε το ότι το θέμα αυτό είναι συστημικό χαρακτήρα στην Ιταλία, το πρόβλημα των μονάδων επεξεργασία. Ήδη τώρα η Ιταλία έχει συρθεί στο δικαστήριο ενώπιον της Επιτροπής τέλο πάντων για τρεις υποθέσεις επί παραβάση. Οπότε και προβλέπουμε στην ολοκλήρωση αυτών των εργασιών για την ε, λίμνη. Έχουμε τώρα τα λοιπάσματα και τα ε, φωσφορούχα γιατί έχουμε μια οδηγία που προβλέπει ότι στην ε, Ήπεθρο των κρατών μελών όταν υπάρχουν υψηλές τιμές ρήπανσης τότε θα πρέπει να αναλαμβάνονται συγκεκριμένε ενέργειες στη ζώνη εκεί που υπάρχουν αυτά τα φωσφορούχα λοιπάζουν να προκαλούν τη ρήπανση. Επομένως είπαμε ότι αυτό που πρέπει τώρα να γίνει είναι να ξεκαθαριστεί γιατί η λίμνη Μπολσένα δεν έχει υπαχθεί σε αυτές τις ε, ευαίσθητες προστατευόμενες ζώνες από τα λοιπάσματα. Έχουμε πάνω στην οδηγία 91 του 271 και θα πρέπει η Επιτροπή να καταλήξει και να κατατάξει εκεί την λίμνη της Μπολσένα. Όταν χαρακτηριστεί μια περιοχή ως ε, ε, ευαίσθητη, τότε λαμβάνονται κάποια μέτρα ούτως ώστε να μειωθούν οι ρήποι από τα λοιπάσματα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα οι βουλευτές. Έχετε το λόγο. Η κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρούνι που ήρθε εδώ για να μας εξηγήσει αυτό το πρόβλημα. Είναι η πολλωστή φορά που αποδεικνύεται ότι στην Ιταλία δεν προσέχουμε πάρα πολύ την σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. Πάρα πολύ συχνά έχουμε μπροστά μας τέτοιες περιπτώσεις. και πολλές φορές μιλούμε για κάποιες τοποθεσίες πάρα πολύ μεγάλη σημασία όπως ε, εν προκειμένου για αυτή την τοποθεσία στο Λάτιο. Είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προστατευτικά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή το 2013. Μας τα εξήγησε ο αναφέρουν. Και θα πρέπει να υποπτεύεται η, η λειτουργία των σκαφών στη λίμνη. Ε, υπάρχουν και θέματα σχετικά με το ψάρεμα που είναι μια δραστηριότητα εκεί. Και έχουμε το 2008 μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Τούσα Και έτσι έχουμε πολλές ενδείξεις που μας οδηγούν στο ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και οι ντόπιοι με επιτροπές τους έχουν αναλάβει ενέργειες και έχουν ζητήσει λύσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτό αφορά και την γεωθερμία της λίμνης. φυσικά και τα ελλείμματα έχουν φρικτές επιπτώσεις. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να περιμένουμε πού θα καταλήξει αυτή η διαδικασία έρευνας και επιπαραβάση. Επομένω, θεωρούμε ότι βρίσκεται ένα δίκο η Ιταλία και αφήνουμε την αναφορά ανοιχτή. Ο κύριο Τσίριο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, αναφέροντα για την παρουσίασή του. Μας εξήγησε και πάλι ένα περίπλοκο πρόβλημα που αυτή τη φορά αφαιρεί μια άλλη βιομηχανία, τη βιομηχανία του τουρισμού. Μιλούμε για υφόρο, βιώσιμο τουρισμό. Πρόκειται για κλάδο της οικονομίας πολύ σημαντικό. Βεβαίως και εδώ πέρα έχουμε σύγκρουση διαφορετικών στοιχείων Έχουμε, όπως είπατε εκεί, κάμπινγκ και άλλες εγκαταστάσεις τουριστικές. Είπαμε ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν αυτές οι επιχειρήσεις τουριστικέ τουριστικές όσον αφορά τα λίματα. Από την άλλη μεριά βέβαια, άμα τις κλείσουν αυτές τις εγκαταστάσεις, τότε και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα έχουμε βέβαια από τη μια μεριά το πρόβλημα το περιβαλλοντικό και από την άλλη το οικονομικό. Δηλαδή στον τουρισμό. Ακόμα δεν έχει καταλήξει η διαδικασία στο ότι υπάρχει η παράβαση, γίνεται η έρευνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σωστό να μείνει ανοιχτή αναφορά. Ευχαριστώ, κύριε Άκεν. Μας σε δύσκολη θέση λίγο αυτό το θέμα. Κάθε φορά που ασχολούμαστε με κάτι που αφορά την Ιταλία, πάντα όλα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα, γιατί η περιβαλλοντικοί νόμοι στην Ιταλία είναι πολύ, πολύ περίπλοκοι. Δεν γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν έχετε λιγότερα χρήματα από εμά. Ίσως έχετε λιγότερους φόρους, ίσως να είναι αυτό ένα πρόβλημα. Και άλλο πρόβλημα είναι η αδιαφάνεια του διοικητικού σας συστήματος. Θυμάμαι και με τα απόβλητα, το Λάτσιο κτλ. Και, και βλέπαμε ότι το μπαλάκι πήγαινε από τον ένα στον άλλον, κανένα δεν ήταν υπεύθυνο. Νομίζω όμως ότι η Ιταλική πολιτική πρέπει να ζητήσουν η Ιταλία να γίνει ένα σοβαρό όριμο κράτος σε ό,τι φορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. ¿Algún, algún diputado más? Άλλος βουλευτής θέλει το λόγο. Όχι. Άρα να ξαναδώσουμε το λόγο στον αναφέροντα. Ε, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Έτσι είναι, για να δείξουν το πρόβλημα όσον αφορά τη γεωθερμία και του κινδύνους. Σύντομα θα είναι αργά. Έχουμε τώρα εκκρεμούσες 22 τουλάχιστον αιτήσει για τη γεωθερμία. Ε, αυτό θα είναι, αυτό θα είναι ένα ε, μια τραγωδία. Τι είναι αυτό, η μαφία, λέει η κυρία Ούκεν. Κοιτάξτε λοιπόν, έχουμε δώσει το λόγο στον αναφέροντα. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει η επιλογή του. Τι θα κάνουμε όσον αφορά την Ελλήνια. Γιατί έχω, όχι τελικά δεν είναι αζωτούχα, είναι, είναι ο φόσφορος αυτό το οποίο βλάπτει την ε, Μπολσένα. Ναι, ναι, ίσως ε, είναι άλλο το στοιχείο, άλλο το υλικό που μολύνει άλλες λίμνες, αλλά για μας εδώ είναι ο φόσφορος. Καλά, λέει ο Πρόεδρος. Σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε, προτείνω να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να διαβιβάσουμε μια επιστολή στις ε, Ιταλικές Αρχές, ούτω ώστε να προχωρήσει, να ξεκαθαριστεί η κατάσταση στην έρευνα τη Επιτροπή. Πάμε στο επόμενο σημείο της ε, διάταξης και είναι η έκθεση Sunset. Είναι Ισπανός, εξ ονόματο της Φουνταθιών ΕΚΟ για παραβίαση της ε, οδηγίας 2008-50 21 Μαΐου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα από το Δήμο Μαδρίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης. Κύριε Νούνιεθ, έχετε το λόγο. Μαρτά Μουνιός Κουέστα. Ε, Καλημέρα σας, λέει. Ναι, ναι, ονομάζομαι Νούνιεθ και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Επιτροπή ή, ή τους αναφέροντες. okay, pues, doy la palabra Alejandro Sánchez. Καλά, τότε να δώσουμε ε, το λόγο στον κύριο Σάντζετ, τον Διευθυντή του Φορέα Φουνταφιών ΕΚΟ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2011 το ΕΚΟ κατήγγειλε στην Επιτροπή σας ότι ο Δήμος Μαντρίτης ε, παραβιάζει την ε, Οδηγεί 2008 κάθετος 50 όσον αφορά την ποιότητα του ομοσφαιρικού αέρα. Μιλούμε για κάποιο είδους σωματίδια που αφορούν το διοξίδιο του αζότου, το όζον και άλλες ουσίες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά αυτά τα σωματίδια, τα αιωρούμενα. στον ονομαζόμενο νότιο διάδρομο της πόλης. Επομένως, πρόκειται για δύο από τις πιο ουσίες, το όζον και το διοξίδιο του αζότου. Πολύ για την υγεία. Έχουμε 20.000 ε, θανάτους ε, στην Ισπανία, 2.000 στη Μαδρίτη. 12 ε, φορές περισσότεροι θάνατοι από όσους από τα τροχεία. Έχουμε επομένως διάφορους οικολόγους, Έχουμε μη κυβερνικές οργανώσεις που είπαν ότι από το 2010-2014 παραδιάστηκαν όλες οι προβλεπόμενες οριακές τιμές και στη Μαδρίτη και αλλού. Και τον Ιανουάριο του 2015 είπαμε ότι σε 6 από του 24 σταθμούς μέτρησης της Μαδρίτης ανέβηκαν οι τιμές πάνω από τι προβλεπόμενες οριακές και αυτό μόνο για πέντε μέρες που μετρήσαν. Οπότε ε, αυτά όσον αφορά το άζωτο αυτή η οδηγία λοιπόν, η 2008 του 50, λέει ότι θα πρέπει να μετράμε τις οριακές τιμές τρία ε, χρόνια συνέχεια. Αλλά εδώ πέρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το 2011 και γι' αυτό και θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απευθεί στην Επιτροπή και να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά δηλαδή το τι έχουν ξεπεραστεί στην Μαδρίτη και γενικότερα στην αυτόνομη περιφερειακή διοίκηση ε, ουρακές τιμές. Πρόκειται για βλάβη στην υγεία των κατοίκων της Μαδρίτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ, λέει Πρόεδρος. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Επιτροπή. Στην κυρία Μουνιώθ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τρία ζητήματα. Πρώτα-πρώτα τα αιρούμενα σωματίδια. Εδώ η κατάσταση έχει προχωρήσει. Και όσον αφορά την παραβίαση των οριακών τιμών έχουμε διαδικασία επί παραβάση. Βρίσκεται εν εξελίξη. 22 Φεβρουαρίου του 2013 απευθύναμε επιστολή στην ε, Ισπανία για παραβίαση των άρθρων 13 και 23 της ε, σχετικής οδηγίας. Απήντησαν οι Ισπανικές αρχές και κατόπιν κάναμε μία μελέτη αυτής της ε, απάντησης και τον Οκτώβριο του 2014 εκδώσαμε τη γνώμη. Απήντησε η Ισπανία και μελετούμε την απάντηση. Υπάρχουν πληροφορίε από κάθε κράτο μέλο για την ποιότητα τη ατμόσφαιρα σύμφωνα με την οδηγία το Σεπτέμβριο κάθε χρονιά. Αυτό είναι το άρθρο 27. Το Σεπτέμβριο του 2014 μα έδωσε η Ισπανία τα στοιχεία που αφορούν το 2013. Αυτέ είναι οι τελευταίε πληροφορίε που μα έστειλε η Ισπανία. Τώρα, όσον αφορά πάντα τα αιωρούμενα σωματίδια από το 2005 έως το 2013 σε πέντε ζώνες μέτρησε τις τιμές και εγκατέσαν και άλλους αθμούς μέτρησες μετά και είπαμε ότι έχουμε υπέρβαση των ορίων σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται. και 2005-2013 στην περιοχή Αστούριας επίσης υπάρχει υπέρβαση των ορίων. Οκτώβριο 2014 είχαμε την τελεγική γνώμη μετά την διαδικασία παραβάση που ξεκίνησε. Έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία επομένως και επί τη βάση αυτών θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τώρα, όσον αφορά το διοξίδιο του αζότου ζητήσαμε διευκρινιστικές παρατηρήσεις από την Ισπανία. Και είπαμε ότι θα πρέπει η Ισπανία να πει πότε θα επαναφέρει τις τιμές στα ωραία που προβλέπονται. Εκεί που τελικά υπάρχει υπέρβαση. Είχαμε υπέρβαση των ορίων από το 2010 στο 2013 στην περιοχή της Βαρκελόνης, στο Λιομπρεγκάτ και στη Μαδρίτη. Και στο ετήσιο όριο και στο ημερήσιο όριο. 10, 11 και 2000 έως το 2013. Αν και έχουμε στοιχεία ε, για τμήμα του 2013, οπότε οι τιμές δεν είχαν υπερβεί τα νόμιμα όρια. ζητήσαμε επομένω να μας, κάνει, να δώσει ευκρινήση η, η Ισπανία και για το τι μέτρα θα λάβει. Τώρα, όσον αφορά το όζον. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά σε σχέση με τα άλλα ρηπαντικά ρηπογόνα στοιχεία. Εδώ έχουμε κάποιες οριακές τιμές που θα πρέπει να οδηγήσουν στη λήψη κάποιων μέτρων. Υπάρχουν κάποιες τιμές στόχοι θα πρέπει να επιστατευτούν όλα τα μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να ληφθούν πάντα στα πλαίσια της αναλογικότητας για τις ζώνες που υπάρχει υπέρβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις επέστρεψα, έπρεπε να βγω έξω, ήταν ε, κάτι επίγον. Με τα χαράς μπορώ να σας πω ότι ο εκπρόσωπος της ε, ο κύριος Νίκολα Μινάση της Ιταλικής Μόνης Αντιπροσωπείας που είχε το ατύχημα ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και είναι εδώ τώρα. Προσπαθεί να λύσει το ζήτημα με την Επιτροπή, με την αναφέρουσα και το συζητούν το θέμα. Μόνο υλικέ ζημιέ δηλαδή στο ατύχημα, αυτό είναι σώο και αυλαβή. Με τα χαρά σα μεταφέρω αυτά τα ευχάριστα νέα. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα ανέφερε για αυτή την αναφορά. Και τώρα να δώσω τα λόγο, no Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομο. <clears throat> Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Και καταρχά να πω ότι η αναφορά αυτή αποδεικνύει το ρόλο που μπορεί να παίξει η Επιτροπή μας. Δηλαδή έχουμε τις καταγγελίες πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και είδαμε από την ίδια τη δραστηριότητα της Επιτροπής ότι ήδη το θέμα αυτό προχωρά. Δηλαδή ότι μετά την αναφορά που έχει έρθει στην Επιτροπή μας και τις καταγγελίες παρατηρούμε ότι και η Επιτροπή έχει ενεργοποιηθεί και έχει απευθύνει συστάσεις προς την ίδια την Ισπανική κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να αναδείξουμε το ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει η δικιά μας Επιτροπή στο ζήτημα αυτό. Επομένως το θέμα της ε, ποιότητας της ατμόσφαιρας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν αφορά μόνο την Ισπανία, αφορά πάρα πολλές χώρες. Να επισημάνω μόνο ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα είχαμε ένα φαινόμενο εθαλομύχλης. Επειδή αυξήθηκε λόγω του, της επιβολής του μνημονίου η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και δεν υπήρχε δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να χρησιμοποιήσουν ε, το καλοριφέρ στις ε, πολυκατοικίες, άρχισαν να χρησιμοποιούν ε, ξύλα και άλλα υλικά προκειμένου να θερμανθούν. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα εθαλομύχλης, το οποίο ήταν πολύ σοβαρό για τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας ε, και τις, ε, που, υπάρχουν και βέβαια να ζητήσουμε την τήρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά διότι πρέπει να παρακολουθήσουμε την υπόθεση όπως έχει παρουσιαστεί στην ε, ίδια την Ισπανία και συγχαίρω τους αναφέροντες για την πρωτοβουλία που έχουν πάρει πάνω στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Now the floor is to you, Rosa. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα ΕΚΟ που ανέδειξε το πρώτο με την αναφορά. Θα πρέπει βεβαίως να μην ανοιχτεί η αναφορά και ακριβώς όπως ε, είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε την διαδικασία παραβάση. Ο Δήμος της Μαδρίτης για το 2008-2011 ε, αποφάσισε να υπάρξουν αυτή η σταθμή μέτρησης ούτως ώστε να ελεγχθεί το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα και από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα με το ε, διοξίδιο του αζότου και έχουμε υπέρβαση των τιμών σε κάποιες τοποθεσίες ακριβώς όπως είπε ο αναφέρον θετικό για την κοινότητα της Μαδρίτης ότι έχουν κάποιο στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας. για να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος 2013-2020. Πάντως για το άζωτο θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουν οι σχετικές μελέτες και επομένως θα πρέπει να δούμε επίσης πού θα καταλήξουν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα ας αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και ας περιμένουμε να δούμε πού θα μα μας οδηγήσει η επικοινωνία μεταξύ Ισπανικών Αρχών και Επιτροπής. Νομίζω ότι η Ρόζα έκανε στην κατάλληλη πρόταση. Πρέπει να μην ανοιχτή αναφορά και να παρακολουθούμε από το συνέγγιστα όσα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που να μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Θα επανέλθουμε. Κύριε Σάντσες, θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που θα κρατήσετε την ε, αναφορά ανοιχτή. Πάντως, σας επισημαίνω ότι η αναφορά είναι ανοιχτή από το 2011 και τώρα έχουμε 15. Και ακόμα ο Δήμος της Μαδρίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κάνανε τίποτα ούτως ώστε να υπάρξει σημαντική μείωση αυτής της ε, ρήπανσης γιατί η Μαδρίτη ε, είναι διαβόητη για το νέφος της σε όλη την Ευρώπη και οι κάτοικοι της Μαδρίτης κάθε μέρα αναπνέουν αυτό το νέφος. Καλά, εντάξει, κάπως μειώθηκε η ατμοσφαιρική ρήπανση λόγω της οικονομικής κρίσης τα δύο τελευταία χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει ε, πιο φράσκα στοιχεία η Επιτροπή, αλλά το 2013 και το 14 και το άζωτο και το όζον έχουν ε, αυξηθεί. Εμείς πάντως θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει με πιο επίγοντα ρυθμό κάτι να κάνει, ούτως ώστε να αναγκάσει τις δημοτικές αρχές της Μαδρίτης κάτι να κάνει. Να σταματήσει τα ωραία λόγια όπως έλεγε το γαλάζιο πρόγραμμα κλπ. Ή κάτι να γίνει τέλο πάντων για την ε, κυκλοφορία των αυτοκινήτων που ρηπαίνει τόσο πολύ. Δεν υπάρχει κανένα αποτελεσματικό μέτρο στη Μαδρίτη που να μειώνει τις συνέπειες από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Και γι' αυτό και έχουμε συνεχή υπέρβαση των ορίων του αζότου. Αλλά και αλλού έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα. Να συγκρατηθούν οι εκπομπές από τους κινητήρες diesel. Κανένα αποτελεσματικό μέσο για την κυκλοφορία για περιορισμό της ταχύτητας ε, στους αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στην πόλη. Οι ειδικοί μας λένε ότι είναι μία από τις βασικές αιτίες της ε, μόλυνσης και της ρήπανσης από το άζωτο. Έχουμε και οικολογικές οργανώσεις που κάνουν ε, μελέτες τελευταία εξαετία. Και είπαν ότι επί τη βάση επισήμων στοιχείων της Διοικητικής Περιφέρειας και του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τα όρια εκπομπών της οδηγίας τα έχουμε υπερβεί. Αλλά θα πρέπει να πιεστούν περισσότερο οι αρχές της Μαδρίτης. Πέρα από μελέτες και καταγγελίες να πιεστούν και από τις ευρωπαϊκές αρχές ούτως ώστε να συμμορφωθούν με τα όσα προβλέπει η οδηγία για την ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει διαδικασία επί Έχει ξεκινήσει. Επομένω, το αφήνουμε ανοιχτό και παρακολουθούμε. Όμω, από περιέργεια, χρειάστηκε να βγω από την αίθουσα. Επομένω, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν διόδια για την είσοδο στην πόλη. Πρόκειται για πρωτεύουσα. Να σα πω ότι στη Στοκχόλμη είχαμε ακόμα και δημοψήφισμα για αυτό το θέμα με όλου του πολίτε. Και είδαμε ότι οι, μισοί κάτοικοι ήταν κατά, η πλειοψηφία ήταν πολύ στενή. Τελικά έχουμε διόδια όμω στη Στοκχόλμη και νομίζω ότι το περιβάλλον η κατάσταση έχει λίγο βελτιωθεί και δεν διαμαρτύρεται ο κόσμο πια. σω πρέπει να γίνει τέτοια εκστρατεία λοιπόν. Κυρία Όκεν, δύο πράγματα. Είχαμε τα ίδια σχέδια και εμείς στην Κοπεχάγη. Δεν υπήρχε πολιτική συνένεση. Επομένως, καταψηφίστηκε η πρόταση του κόμματό μου. Συμφωνώ πολύ με εσά, αλλά να, να πω... Η πρώτη αναφορά που είχα εξετάσει το 2007-2008 ήταν για τον M30. Ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος στη Μαδρίτη. που είχε γίνει χωρίς ε, πρώτερους ελέγχους ή μελέτες. Δεν είχαν καν εξετάσει τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές της Μαδρίτης προσπάθησαν να, ε, να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αποκαλώντας το ΚΑΓΕ, έναν απλό δρόμο δηλαδή, τον αυτοκινητόδρομο. Συμφωνώ όμως με την πρόταση για τα διόδια. Γιατί θυμάμαι πως ε, είχαμε αντιμετωπίσει την κατάσταση τότε και νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Πρόεδρος, ε, σας διαβεβαιώ ότι θα εξακολουθούμε να προσέχουμε και να παρακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Όμως, ίσως πρέπει να αρχίσετε και εσείς να κάνετε πιο έντονες εκστρατείες ε, στη χώρα σας σας εύχομαι καλή επιτυχία. Φτάνουμε στο τέλος των εργασιών για σήμερα το πρωί. Είστε ελεύθεροι τώρα να κάνετε τα τηλέφωνά σας, να δείτε τα mail σας, κάποια στιγμή να φάτε και το μεσημέρι και θα τα πούμε στις 3 με τον Επίτροπο Τίμερμαντς. Τα λέμε τότε λοιπόν.